Άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Je voudrais m'assurer que l'ordre du jour... Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται λοιπόν το σχέδιο ημερήσιας διάταξη. Έχετε λάβει τα πρακτικά της 3ης Απριλίου. Ελάβατε γνώση αυτών. Παρατηρήσεις, σχόλια. Αν όχι, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και φτάσαμε στις ψηφοφορίες. Πρώτη έκθεση που να ψηφίσουμε. Η κυρία Τωμά, χωρίς μικρόφωνο, δεν έχετε την κάρτα σας. Très bien. Donc, lorsque... Μάλιστα. Κατά τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, λοιπόν, όταν ανακοινώνω το αποτέλεσμα... Θα σας παρακαλέσω να μας λέτε τι ψηφίζετε κάθε φορά. Για να μην νιώσετε την απογοήτευση ότι δεν θα ληφθεί η ψήφο σας υπόψη. Μαθαίνω ότι είχαμε προβλέψει να ψηφίσουμε στις 11 παρατέταρτο λέει και είναι παρά 20. Δεν ξέρω, έχετε κανένα τραγουδάκι να μας πείτε, λέει ο πρόεδρος. Ένα παραμύθι. Έχει η κυρία Τωμά να φέρει την κάρτα της, ορίστε. Ναι, <laughs> ναι, on peut l'applaudir, parce que vraiment... Donc la séance... χειροκροτά. Λοιπόν, πέντε λεπτά διάλειμμα. Rappelle-toi, Barbara, Bonjour Paul.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 which, which says that the Court of Auditors has to come with a special report. Madame Thomas est de retour, il est donc euh, 10h40. Επέστρεψε η κυρία Τωμά και πήγε και η ώρα 11 παρατέταρτο, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Nous abordons la séquence des votes. Ώρα ψηφοφορίας λοιπόν. Η πρώτη έκθεση είναι του κυρίου Σαρβαμά για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έχετε τις κάρτες σας στα μηχανήματα όλοι παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, 32 αναμένεται να ψηφίσουν. Κάποιος καταψήφισε τη δοκιμαστική. Τροπολογία υπάρχουν δύο ψήφοι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπάρχουν τρία υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Η πέντε υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 14 καταπίπτει η τροπολογία υπερθμών ένα ψηφί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Επόμενη έκθεση. Είναι έκθεση του κυρίου Όλμπριχτ. Με θέμα την ενίσχυση συμμετοχής των εταίρων και της προβολής της επιδόσης των Ευρωπαϊκών Διαρθωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Τροπολογία παρθμόν 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Την τροπολογία παρελθόν δύο ψηφίσμα. Πέρας. Απορρίπτεται. 20-12. Η τροπολογία υπάρχουν 3. πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπάρχουν 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνόλου του κειμένου ηλεκτρονικά αρχής ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. 30 υπέρ, 3 κατά συγχαρητήρια κυρία Όρμπριχτς. Και τώρα έχουμε την έκθεση του κυρίου Ντεπχέ με θέμα τη μετανάστευση και το Δουβλίνο. Είναι σχέδιο γνωμοδότησης. Το κύριο Ντεπχέ για την αναθεώρηση ε, του κανονισμού του Δουβλίνου. Μία βουλευτής έχει κάνει 500 τροπολογίες. Η κυρία Μοντέλ, η οποία διακρίνεται έτσι. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Από την προηγούμενη ψηφοφορία. Μπορεί να εμφανιστεί και κάποια μέρα να μας εξηγήσει γιατί κάνει τόσο πολλές τροπολογίες βασικά διαγραφή ζητάει το κειμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μη τροποποιημένων ε, ε, παραγράφων που δεν αφορά η αναδιατύπωση. Η γραμματεία ε, μας ζητάει να τα ψηφίσουμε όλα αυτά μαζί. Θέλει κανείς το λόγο. Κύριε Τζάνη, παρακαλώ για αυτή την υπόθεση. Καταρχάς ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους γιατί είναι μια πρακτική την οποία δεν συμμερίζομαι. Δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία ήταν 15 Φεβρουαρίου. Είχα συζητήσει με τη συνάδελφο και έτσι ώστε να μην συμβούν πλέον τέτοιου είδους ε, ε, ε, πράγματα, γιατί είναι λυπηρό αλλά και ενοχλητικό. Θα είναι η τελευταία φορά ε, που, θα, που γίνεται αυτό το πράγμα και αυτός ο τρόπος εργασίας της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που επαναφέρετε την κυρία Μοντέλ σε μια πιο υπεύθυνη ε, στάση και πιο ε, με πιο σεβασμό να δείχνουν στους συναδέλφους γιατί αυτό το πράγμα είναι παρενόχληση. Ε, ωραία. Έχουμε λοιπόν υπό το 174 αναθεωρημένο μπορούμε να θέσουμε unblock σε ψηφοφορία μια σειρά ε, τροπολογιών εκτός εάν ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία από μια ομάδα ε, πολιτική ή από τουλάχιστον τρεις βουλευτές. Ακόμα και αν σε περίπτωση που ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία μπορώ να αποφασίσω μετά από την απόρριψη ενός κάποια, μιας κάποιας τροπολογίας να βάλω unblock ε, σε ψηφοφορία ε, άλλες τροπολογίες που έχουν περιεχόμενο ή ε, παρόμοιο ή στόχους παρόμοιους. Δεν νομίζω να υπάρχει αντίρρηση λοιπόν να προχωρήσουμε έτσι και να ψηφίσουμε unblock. Επίσης να σας θυμίσω ότι όσον αφορά το άρθρο 154 αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω πως έχουμε ρυθμίσει το ζήτημα και ο κύριος Τζάνι αυτό μας είπε ότι δεν θα ξαναγίνει, δεν θα επαναληφθεί, οπότε θα ψηφίσουμε unblock. Ε, λοιπόν, τροπολογίες 93 μέχρι 554 που περιλαμβάνονται και περιγράφονται στη σελίδα 1 μέχρι και 22 του καταλόγου ψηφοφορίας σας. Συμφωνείτε αγαπητοί συνάδελφοι να απορρίψουμε αν όλες αυτές τις τροπολογίες, δηλαδή 22 πρώτες σελίδες του καταλόγου ψηφοφοριών μας. Ποιοι είναι υπέρ της απόρριψης αυτών των τροπολογιών. Παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι όσοι είστε υπέρ της κατάρρευσης, της απόρριψης. Μάλιστα, ευχαριστώ. Υπέρ της διατήρησης, κανείς. Αποχές, όχι. Ωραία. Το εκτιμώ πάρα πολύ ε, αυτή την ομόφωνη θέση της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Και τώρα θα ψηφίσουμε άλλες τροπολογίες, μια σειρά, ορισμένες εκ των οποίων είναι της κυρίας Μοντέλ, αλλά που δεν ήταν ε, μέσα στις πρώτες ε, ψηφοφορίες που κάναμε έναν μπλοκ, 112 λοιπόν, υπέρ, κατά, Αποχές ε, απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα, συμβιβαστική 3 Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται. Στο le 3. Πέρας. Πέρας. Je m'en Εγκρίνεται. 29 έναντι 2 και 2 αποχές. 398 υπερκατά κατά, αποχές απορρίπτεται. 400 υπερκατά αποχές απορρίπτεται. 401 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. On va voter à main levée. Qui est pour Qui est contre Υπέρ κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Και contre. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 415. Ε, Υπέρ. Α, όχι, έχει καταπέσει, μάλιστα. Συγγνώμη. 417. 417. Oui, il tombera si. Donc le 417 qui est pour. 417 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 420 είχε το, το ίδιο αντικείμενο απορρίπτεται το 11 και το 419, ή 11 μάλλον και το 419 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. 421 και 422 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 έχει καταπέσει επειδή εγκρίθηκαν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 παρότι κρίθηκε το 6 δεν καταπέπτει 4, η 7 υπέρ κατά αποχές ε, ε, εγκρίνεται. 410 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συγγνώμη, ε, διορθώνει ο πρόεδρος εγκρίνεται. 453 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται. Scrutin Πέρας. Πέρασε. par 20 voix contre 12. 33 έναντι 12 ε, απορρίπτεται. Συγγνώμη, 23 έναντι 12 απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια σας. Λοιπόν, τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 14 est adopté par 20 voix contre 13. Εγκρίνεται 21 έναντι 13. Τροπολογία 15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 532. Υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται. 534. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα προτείνω ψηφοφορία unblock για τα εκτιμώντας. Πρόκειται για τις τροπολογίες της κυρίας Μοντέλ. Για το σύνολο των τροπολογιών της κυρίας Μοντέλ, δηλαδή οι σελίδες 25 και 26 του καταλόγου ψηφοφορίας, ποιοι είναι υπέρ. Contre. Κατά. Αποχές απορρίπτονται και ξανασυνεχίζουμε με τις τροπολογίες επί των ε, θεολογικών ε, σκέψεων, τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 ε, ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές ε, γκριν, ε, απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του κυρίου Ντεπρέ υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 έχει καταπέσει, η 47 επίσης, η 3 ναι, καταπίπτει, η 52 Α, η 3, συγγνώμη. Να το ψηφίσουμε πρέπει. Τροπολογία 3. Υπέρ της ε, τροπολογίας 3, υπέρ κατά αποχές ε, γκρίνεται. Τροπολογία 52 καταπίπτει γιατί υπερψηφίστηκε το 3. Η 3 55, 58, 61 και 63 έχουν το ίδιο δικείμενο και τις ψηφίζουμε από κοινού. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 καταπίπτει. 59 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται.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 μια μεταφορά πιστώσεων ω αποτέλεσμα των εκθέσεων που ψηφίσατε για την έκθεση του κ. Σαρβάμα για μεταφορά 2.641.800 ε, ευρώ για την υπόθεση της Νόκια, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 19 υπέρ, μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Για τον κύριο Τάχον δεν υπάρχει κάποια αίτημα μεταφοράς πιστώσεων, ούτε από την κυρία Χολμάγερ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως θα μπορούσε στην επόμενη συνεδρίαση να μας υποβάλει μια έκθεση σχετικά με τα κτίρια ΙΠΑ και ΙΜΑ, γιατί ε, είναι υποθέσεις που διαρκούν πολύ. Για το ΙΜΑ δεν έχει γίνει αποδεκτό μάλλον, γιατί δεν είχαμε break-up clause. Θα θυμάστε ότι είχαμε εκφράσει την ε, ε, γνωμοδότησή μας Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει άλλο σημείο στο Λονδίνο ή σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία που να μπορούσε να μπει εκτός από το σύντη του Λονδίνου. Είχαμε πει ότι δεν υπάρχει break-up clause. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο διαφορετικό σενάριο. Πάντως, επειδή μιλάμε για πολλά χρήματα και για το ΕΠΑ και για το ΕΜΑ, θα θέλαμε από την Επιτροπή κάποια ενημέρωση. Δεν ξέρω σε σχέση με το Brexit, μήπως ε, αλλάζουν τα πράγματα. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit σίγουρα θα αναφερθεί το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας απαντήσει τώρα, φαντάζομαι δεν θα μπορεί τώρα, πάντως διατυπώσαμε το ερώτημα και θα περιμένουμε απάντηση από την Επιτροπή σε κάποια επόμενη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δίνουμε το λόγο στην Έντερ Ζαμπάλ που θα μας μιλήσει για τον τριμερή διάλογο για το Ταμείο και τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, μπαίνουμε τώρα στη φάση των τριμερών διαλόγων λίγες εβδομάδες. Δεν ξέρω από πότε συζητάμε αυτή την έκθεση. Τρεις φορές συνεδριάσαμε σε τριμερή διάλογο και η αλήθεια είναι ότι προκολαράμε καλά με σταθερά βήματα και θα συμφωνήσουμε για σημαντικά θέματα. Κάποια στιγμή καθορίσαμε εννέα σημαντικά θέματα που θέλαμε να διαπραγματευτούμε για τις δύο αυτές εκθέσεις. Και βέβαια μετά κοιτάξαμε όλες τις τροπολογίες. Εννέα λοιπόν είναι τα θέματα. Τέσσερα από τα οποία έχουν ήδη κλείσει Υπάρχει μια προσυμφωνία και περιμένουμε την οριστική. Είναι όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολιτική ισότητας, κλιματική αλλαγή και ευελιξία και μεταφορά πιστώσεων ε, που δεν έχουν απορροφηθεί. Αυτά έχουν σχεδόν κλείσει και περιμένουν την τελική συμφωνία. Υπάρχουν δύο θέματα αρκετά σημαντικά, το ένα τουλάχιστον, που σχεδόν έχει κλείσει και την επόμενη φορά θα οριστικοποιηθεί και θα συμφωνήσουμε. Το ένα είναι ε, ό,τι έχει να κάνει με το reporting, τη διαφάνεια και την απόδοση λογαριασμών. Τα τρία θεσμικά όργανα συνεννοούμαστε για να δούμε πώς μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε και να εξασφαλίσουμε εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Έχουμε εξηγήσει όμως στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εδώ έχουμε και κανόνες και αναγνωστήρια και μπορούμε να κινητοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί ε, ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των διαβαθμισμένων εγγράφων ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων που μπορεί να έχουμε εμπορικό απόρριτο, ευαίσθητες πληροφορίες και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία εξίσου ε, ευαίσθητα, αλλά και τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ε, μια διαβίβαση, ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει, να δούμε με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα γίνει αυτό. Και το θέμα της φορολογίας, που πιστεύω θα συμφωνήσουμε πλέον, ήδη από τώρα ξέρουμε ότι το Συμβούλιο εκπονεί μια πρόταση βάσει των όσων προτείναμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα. Αλλά θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι και η Προεδρία και το Συμβούλιο γενικά, παρά την κάποια διστακτικότητα στην αρχή, στις διαπραγματεύσεις έδειξαν πολύ ανοιχτή στάση και συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει πρόοδος η φορολογία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη φορολογική απάτη, φοροαποφυγή, τις επιθετικές φορολογικές ε, συμφωνίες, τα περίφημα rulings κτλ. Και πώς δρούν κάποιες χώρες ως διαμεσολαβητές για να γίνονται κάποιες σκοτεινές ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Εκεί μας λείπουν κάποιες λεπτομέρειες τελικές όμως και θα συμφωνήσουμε πιστεύω και θα είναι σημαντικότερη φορολογική συμφωνία τουλάχιστον μέχρι τώρα για τα φορολογικά θέματα μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτά. Τρία θέματα εκκρεμούν ουσιαστικά ανοιχτά. Το ένα έχει να κάνει με μια καταξισοδότηση πράξη για την τροποποίηση του παραρτήματος παριθμών 4 και αυτό ε, έχει να κάνει με τις πολιτικές που θα διέπουν την εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, αναζητούμε έναν τρόπο να επικαιροποιούμε αυτό το παράρτημα χωρίς να ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου ε, ολόκληρης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν γίνεται να το κάνουμε αυτό χωρίς κατεξοδότηση πράξη θα συμφωνήσουμε. Αυτό είναι σχετικά ίσονο σημασία. Τα δύο σημαντικότερα τώρα που εκκρεμούν είναι η διαχείριση του Ταμείου, πρώτα, γνωρίζετε ότι Κομισιόν και Κοινοβούλιο προτείναμε να ανατεθεί η διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους αποτελεσματικότητας, για λόγους οικονομίας και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται άλλα αντίστοιχα ταμεία και ξέρει και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Πλην όμως τα κράτη-μέλη αρνούνται κατηγορηματικά να ε, δώσουν τη διαχείριση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το θέμα παραμένει έτσι σε παράλυση. Και ομολογώ ότι με εκπλήσει πολύ αυτή η στάση του Συμβουλίου. Διότι έχει αποδεχθεί περίτρανα και από έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι εξοικονομούμε χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δωρεάν θα έρθει να διαχειριστεί αυτό το ταμείο. Δηλαδή, δεν έχουμε καθόλου συμπληρωματικό κόστος. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα την πληρώνουμε και όλα σε αυτή την υπηρεσία. Τι είναι αυτό, εξωτερήκευση μια δουλειά που μπορεί να γίνει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό είναι χρηστή οικονομική διαχείριση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Συνεπώς όταν διαρριγνύει τα ημάτια του το Συμβούλιο για ε, προϋπολογισμό βάση αποτελεσμάτων και χρηστή διαχείριση και όχι κατασπατάληση και ξέρω εγώ τι. Και το τελευταίο θέμα που εκκρεμεί, όπως το ξέραμε από την αρχή, είναι τα ποσά και οι οροφές. για την εξωτερική εντολή της ΕΤΕΠ. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει αύξηση, το Κοινοβούλιο ζήτησε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση για να αντισταθμίζεται αυτή η προκαταβολή, μια δαπάνη που είχε γίνει σε χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, αλλά το Συμβούλιο δυνατή να κινηθεί. Ξέρουμε, όταν πρόκειται για δημοσιονομικές συζητήσεις με το Συμβούλιο, χαιρετίσματα. Και μέχρι τώρα τα έχει στυλώσει. Και όσο έτρεχαν οι διαπραγματεύσεις, ε, μάθαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε να αφαιρεθεί το θέμα αυτό από την ημερησία διάταξη. Ε, οι δύο τελευταίοι διάλογοι έγιναν την Πέμπτη και τη Δευτέρα που μας πέρασε και ρώτησα το Συμβούλιο αν είναι διαθέσιμο ή αν θεωρεί σκόπιμο να δω πώς να το διατυπώσω τώρα να γίνει το εξή. Να μην λάβουμε τώρα απόφαση οριστική αύξηση του ποσού ε, της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕΠ, αλλά να το συνδέσουμε με ένα προαπαιτούμενο. Αν υπάρχουν πιστώσεις διαθέσιμες στα επόμενα δημοσιονομικά έτη. Με ποια έννοια. Ο στόχος να παραμείνει με ο ίδιος, πλην όμως Το Συμβουλίο δεν χρειάζεται να το αποφασίσει τώρα, αλλά χρόνο με το χρόνο πώς ε, εκτελείται ο προϋπολογισμός και αν από την κατηγορία 4 περισσεύουν λεφτά, να μπορούμε να τροφοδοτούμε αυτό το ταμείο για να αυξηθούν οι πιστώσεις. Είπα στο Συμβούλιο ότι αυτή η πρόταση είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο για να βολιδοσκοπήσει η Προεδρία αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο συμφωνίας. Να τα βρούμε κάπου στη μέση δηλαδή. Όχι στα ποσά επαναλαμβάνω, αλλά στο χρόνο τουλάχιστον. Με προς στιγμή το Συμβούλιο ε, αγρό αγοράζει. Θα το κοιτάξουν, λέει, να το κοιτάξουμε και εμείς όμως ε, προσεκτικά πώς μπορούμε τεχνικά και νομικά να προσαρμόσουμε αυτή την πρόταση. Με τη βοήθεια των δικών μας υπηρεσιών και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά εδώ και προσπαθεί να φέρνει κείμενα για να συγκεράσει τις απόψεις ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αλλά όπως είπα και στο Συμβουλίο και τους εξήγησα, η πρόταση αυτή είναι όχι τόσο πολιτική, αλλά είναι μια βολιδοσκόπηση, επαναλαμβάνω, του Συμβουλίου για να δούμε τις προθέσεις τους. Τις επόμενες εβδομάδες ε, υποθέτω ότι θα έχουμε συνομιλίες με Κομισιόν και Συμβούλιο. Γιατί δυστυχώ μέχρι 30 Μαΐου δεν έχουμε άλλη συνεδρίαση ε, διαλόγου. διαλόγου, Μεσολαβή Στρασβούργο, Τυρκουάς Εβδομάδα και πάει λέγοντας. Αυτά. Άτυπε, συζητήσει και επαφέ θα έχουμε για να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε και να οριστοκοπήσουμε τις ε, διαπραγματεύσει στι 30 του μηνό. Νομίζω ότι σα τα είπα όλα. Αυτά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Euh, Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γκαρδιαζαμπάλ που μα, ε, τα εξήγησε όλα. σα ε, παρακολουθούμε. παρακολουθούμε την ένταση με την οποία ασχολήσαμε τον τριμερή διάλογο για το Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θα παρακολουθούμε τι πρόοδου που γίνονται για να ασχοληθούμε και με τα μη συνεργάσιμα κράτη, με προλογικούς παραδείσους, με ε, χώρες που μπορούν να χρησιμεύσουν για αποφυγή ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην παραλείψει κανένα θέμα σε αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρατε τρία θέματα για τι ε, εξουσιοδότηση πράξη, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Για ε, τη διαχείριση ε, κονδυλίων νομίζω ότι μιλάμε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Θα έπρεπε να ξέρουμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σε σχέση με τις ε, ε, ικανότητες της, ε, με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Να είναι ξεκάθαρο και να μην υπάρχει αμφιβολία. Για το τρίτο θέμα που αναφέρετε, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να προσαρμόσουμε όσο περνάει ο καιρός. Ο κύριος Δεπχέ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Και εγώ θεωρητικά είμαι μέλο τη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, αλλά δυστυχώ μόνο σε μία συνεδρίαση του τριμερού διαλόγου μπόρεσα να είμαι παρόν. Εκφράζω την πλήρη ε, υποστήριξή μου στην ΕΝΤΕΡ για την εξυπνάδα και την αποφασιστικότητά τη κατά τι διαπραγματεύσει. Ένα πολύ μικρό πρόβλημα υπήρξε που ήταν διαδικαστικό όσον αφορά την ε, δυνατότητα αύξησης του διαθέσιμου ποσού. Όσον αφορά τη διαδικασία, δεν έγιναν ε, οι διαβουλεύσεις όπως θα έπρεπε. Όμως, επί της ουσίας, συμφωνούμε απολύτως με, τη θέση, με την πρότασή της και υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της και θα την υποστηρίξουμε κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ο κ. Κέρμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Εντέρη για την προσπάθειά της και για την ένταση με την οποία λιονταρίσια ανταπεξέρχεται στις διαπραγματεύσεις. Δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε τα σωστά επιχειρήματα όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεκπεραιώνει αυτά τα θέματα και δεν, έχουμε, δεν σημαίνει τα πάνες για μας. Ίσως δεν είναι σωστό το επιχείρημα. Ε, διότι υπάρχουν δαπάνες. Το θέμα είναι αν οι δαπάνες αυτές δίδονται από κάποιον άλλον, διότι το αναθέτουμε σε κάποιον εξωτερικό, ή αν ε, χρησιμοποιούμε ε, δικό μας προσωπικό. Πάντως η χρηματοδότηση δίδεται ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι ποιος θα το κάνει καλύτερα και ποιος θα το κάνει πιο αποτελεσματικά. Δηλαδή, λέει ο Πρόεδρος διακόπτοντας, μήπως εννοείται ότι η Επιτροπή έχει πάρα πολλούς υπαλλήλους, υπερβολικά πολλούς. Ίσως και να εννοώ και αυτό, αλλά δεν έλεγα ακριβώς ε, αυτό. Αλλά όντω, όταν σκεφτόμαστε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, είπαμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ασχοληθεί. Τώρα, όταν μιλάμε για ένα νέο ταμείο, το οποίο έχει μια παρόμοια δομή, ίσως και για αυτό το θέμα, ίσως να υπάρχει κάποια ανάθεση καθηκόντων από την ε, ΕΤΕΠ ή από την Παγκόσμια Τράπεζα. Δεν έχω αντίρρηση να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ε, πιστεύω ότι είναι λάθος η αρχική διατύπωση ότι είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα, όσον αφορά το Ταμείο Επενδύσεων, το Ταμείο Εγγύησεων, για επενδύσεις στην Αφρική ε, είναι ένα μέσο χρήσιμο και λογικό, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων. Γιατί νομίζω ότι εδώ έχουμε δύο διαφορετικές παραμέτρους. Το Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων έχει ένα πρόβλημα προσθετικότητας και υπάρχει και ένα πρόβλημα όσον αφορά τους κινδύνους αυτό ε, στην περίπτωση της Αφρικής θα έχουμε ε, ισχύει το αντίθετο, δηλαδή ε, θα υπάρχει μικρότερο πρόβλημα προσθετικότητας και μεγαλύτερο πρόβλημα κινδύνων. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση κινδύνων. Και θα πρέπει να προσέξουμε οι τρεις πυλώνες για την βοήθεια προς την Αφρική αλλά και για τις ε, χώρες ε, της γειτονίας θα πρέπει να ε, υπάρχουν και οι τρεις πυλώνες, να μην ξεχνάμε το δεύτερο και το τρίτο. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν επιτόπου οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνουν βιώσιμες επενδύσεις. Τέλος, πιστεύω ότι και εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια και τα κονδύλια τα οποία δίδουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσουν παράγοντα μόχλευσης για μεγαλύτερες επενδύσεις και αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο, το ο Πρόεδρος. Να ζητήσω από την Έντα να, κάνει, να μας δώσει τα συμπεράσματα. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Κέλμελ ρώτησε ε, αν είναι δωρεάν οι υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα γι' αυτό είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται ήδη ε, τέτοιου είδους προγράμματα και ενεργητικά και έχει ειδική ομάδα που ασχολείται με αυτά. Δηλαδή το να προσθέσουμε άλλο ένα ταμείο δεν επιβαρύνει οικονομικά δεν θα προσλάβει υπαλλήλου. Δεν αυξάνεται το κόστος. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πληρώνουμε την υπηρεσία αυτή. Είναι καθαρή οικονομία αυτό που κάνουμε. Και τα χρήματα αυτά που θα εξοικονομήσουμε θα παραμείνουν στο Ταμείο ε, για τις ανάγκες του Ταμείου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλού, σε δράσεις, σε έργα και όχι σε λειτουργικό κόστος. για να χρηματοδοτούμε επενδύσεις στο εξωτερικό. Είναι απόλυτη οικονομία, καθαρή οικονομία. Το είπε και ο κύριος Αχτουή. Και για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για τα ίδια πρόκειται. Άλλο είναι η διαχείριση του ενεργητικού του ταμείου που είναι οικονομική, χρηματοοικονομική και άλλο είναι ποιος εγκρίνει τα προγράμματα, ποιος αποφασίζει, ποιος τα αξιολογεί. Και στο ΕΦΣΙ και εδώ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παίρνει τις αποφάσεις ε, για τα έργα. Το θέμα είναι ποιος κάνει τη λογιστική δουλειά, την οικονομική. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τελείως διαφορετικά. Αυτά. Eh Θα διακόψουμε τώρα και θα ξαναρχίσουμε στις 12 το μεσημέρι, γιατί τότε έχουμε προγραμματίσει κοινή συνεδρίαση. Ε, Μπάτζ. Λυπούμε, ναι, τελείωσαμε λίγο πολύ γρήγορα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το δεχτήκατε κι εσείς ότι ήσασταν σύντομοι. Λοιπόν, ε, διακόπτουμε μέχρι τις 12.